Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή, η αρχή της επικουρικότητας και η καθολικότητα των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συντάκτες που θα πάρουν το λόγο. Πρώτος ο κύριος Όλμπριτς για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η προφορική αυτή ερώτηση που έχουμε υποβάλει ήταν απόρρια μιας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκίνησε από την επιλεξιμότητα και ποιος ήταν δικαιούχος κοινωνικής στέγης στην Ολλανδία. Ε, και τελικά κατέληξε το Κοινοβούλιο γιατί έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και σημαντικές. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν διαφορετικοί ορισμοί της κοινωνικής στέγης ε, των εργατικών κατοικιών ε, και κατά πόσο είναι κοινοφελής υπηρεσία και παροχή των συστημάτων Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια λοιπόν από χώρα σε χώρα ε, και για το ποιο δικαιούται ε, την κοινωνική στέγη αλλά και ποιος ε, διαχειρίζεται τη στέγη αυτή και ποιο τη χορηγεί. Σε άλλες χώρες είναι το δημόσιο, σε άλλες χώρες είναι ιδιωτικοί οργανισμοί. Η συζήτηση αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική και ε, αφορά και την Ευρώπη διότι ε, τίθεται ζήτημα διαρθρωτικό ταμείο. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μία και μόνη ε, ρύθμιση, ένας ορισμός για τις ε, κοινωνικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την κοινωνική κατοικία. Θα ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ελάχιστο εισόδημα ε, της οικογένειας του νοικοκυριού όπως το κάνει ε, η Ολλανδία για παράδειγμα. Συντάκτη για, για τρία λεπτά κυρία Ρούλε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για μια δήλωση τύπου που δημοψήφισε στις 19 Δεκεμβρίου του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την απόφαση αυτή για την ενίσχυση το σύστημα ε, της ε, Ολλανδικής Κοινωνικής ε, Κατοικίας. Και παραθέτω, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικυρώνει τη μέχρι τώρα πολιτική ότι τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλο περιθώριο ρηγμών όταν ορίζουν τα κριτήρια και τα ισχύοντα για τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και γενικού κοινωνικού συμφέροντος. Και ρωτώ τώρα, πώς ταιριάζει αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη νέα. Είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό πώς ε, ορίζεται με την αναλογικότητα και με την επικορικότητα και πώς σχετίζεται με αυτές τις δύο αρχές. Μπορεί τυπικά να αναγνωρίζεται ένα κοινωνικό μείγμα για την ανάγκη αυτή, αλλά υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις και ταυτόχρονα ε, ορίζεται 10% ε, πάνω από το κατόφλι των 30.000 ε, ευρώ. Και ε, λέγουν επίσης ότι κάποια στιγμή μπορεί να αυξηθεί και το 10% για κριτήριο κοινωνικής στέγης. Και μετά θα πρέπει αυτό να αντισταθμιστεί με συμψηφισμό στο εσωτερικό της χώρας. Είναι πάρα πολύ άκαμπτη λοιπόν αυτή η ρύθμιση και δεν καταλαβαίνω πώς συνδέεται με τα προηγούμενα και με την επικουρικότητα και το δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν ε, αυτά τα ζητήματα, να αποφασίζουν με μεγάλο περιθώριο ελιγμών, όπως είπε τότε ε, το Δεκέμβριο στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρούλε. Τώρα άλλη συντάκτης, η κυρία Καστέκ, για δύο λεπτά επίσης. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Στρέφομαι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτή την κοινοποίηση για την βοήθεια σε σχέση με τις κοινωνικές ε, κατοικίες και συγκεκριμένα τις κατοχώρες όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ευθυγράμμιση με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Αντί λοιπόν να ζητήσει την, σε βάθος μεταρρύθμιση ε, του τομέα αυτού και των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος θεωρώ ότι έχει ερμηνεύσει και ορίσει περιοριστικά τις υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος. Η Επιτροπή αναγνωρίζει βέβαια τον κοινωνικό χαρακτήρα των δημόσιων υπηρεσιών, ωστόσο τονίζει ότι θα πρέπει να ορίζεται και παραπέμπω σε αυτά που λέτε σε άμεση σχέση με τις ε, μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες. Επομένως η προσφορά κοινωνικών κατοικιών στην ε, Ολλανδία ήταν υπέρ αυτών ουσιαστικά για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ε, των ε, μειονεκτικών ομάδων. Η πρόταση μεταρρύθμισης του τομέα αυτού που προτείνει η Ολλανδική κυβέρνηση περιορίζει στο 10% τον όγκο των κοινωνικών κατοικιών που μπορούν να δοθούν σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πάντοτε όμως με βάση κοινωνικά κριτήρια και κατά σειρά προτεραιότητας. Αυτός ο περιορισμός ουσιαστικά θέτει εκ νέου αφισβήτηση μια άλλη αποστολή τη δημοσία υπηρεσία που πληρεί ακριβώ η υπηρεσία δημόσιων ε, κοινωνικών ε, κατοικιών, που είναι ουσιαστικά η αστική και κοινωνική ανάμειξη κατά κάποιο τρόπο, όπως ορίζεται και από τον Ολλανδό νομοθέτη. Επομένως, το θέμα το οποίο με αφορά είναι το εξή. Με ποια νομική βάση τη συνθήκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να θέσει αμφισβήτηση τον καθολικό χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών και με ποια νομική βάση μπορεί να επιβάλλει σε ένα κράτος μέλος να επαναπροσδιορίσει την αποστολή που έχει ε, θεωρήσει ότι πληρεί μια τέτοια υπηρεσία. Ευχαριστώ. Τώρα, εξ ονομάτου της Επιτροπής, ο κύριος Άντορο Επίτροπος έχει το λόγο. Uh, Κυρία Πρόεδρε, ε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, ε, για τις ερωτήσεις που τέθηκαν, πρώτα απ' όλα η Κομισιόν πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός για την κοινωνική κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της καθολικότητας, και, δεύτερον, και τρίτον για το όριο εισοδήματο για την πρόσβαση στην κοινωνική κατοικία. Πριν απαντήσω στι ερωτήσει αυτέ, πρέπει να σα πω ότι αποδίδει μεγάλη σημασία η Κομισιόν στην κοινωνική κατοικία, που είναι ένα βασικό εργαλείο για τι πολιτικέ κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τι ερωτήσει 1 και 2, θέλω να είμαι απολύτω σαφή. Η Κομισιόν δεν επιβάλλει έναν ενιαίο ε, ορισμό για την κοινωνική κατοικία και σέβεται πλήρω την αρχή τη επικουρικότητα. Οι κύριοι Ευρωβουλευτέ πολύ σωστά αναφέρθηκαν στην απόφαση τη Επιτροπή του 2005 για κρατικέ ε, επιχορηγήσει για υπηρεσίε γενικού ε, ε, ενδιαφέροντο. Η απόφαση αυτή παρέχει ασφάλεια δικαίου για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι ενισχύσεις για την κοινωνική κατοικία έχουν προτιμησιακή μεταχείριση, διότι εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίηση ανεξάρτητα από τα ποσά τα οποία εμπλέκονται. Σύμφωνα με την ε, απόφαση αυτή, η εξαίρεση αυτή ισχύει όταν η κοινωνική κατοικία είναι, ε, ε χαρακτηρίζεται σαν υπηρεσία γενικού ε, δημοσίου ενδιαφέροντο από το ίδιο το κράτο μέλο, Ούτω ώστε να συμφωνεί ο ορισμό αυτό σύμφωνα με τις παραδόσεις του κράτου σχετικά με τι κοινωνικέ παρεμβάσει. Επίσης υπάρχουν οι ανακοινώσει τη Κομισιόν του 2006 και του 2007 που τονίζουν την ε, υπευθυνότητα και τη διακριτική ευχέρεια ε, του κράτους μέλους όσον αφορά τον καθορισμό των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, πιο πρόσφατα, αυτό υπογραμμίστηκε στο σχετικό πρωτόκολλο. Όμως, Εφόσον μιλάμε για κοινωνική κατοικία, δεν μιλάμε γενικώ για στέγη, αλλά για στέγη που παράγεται με βάση κοινωνικά κριτήρια. Γι' αυτό υπάρχουν τα εκτιμώντα στις αποφάσεις, στην ε, απόφαση του 2005 που αναφέρεται ε, σε πολίτες σε βρισκόμενους σε μικρική θέση ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που λόγω ε, κοινωνικών περιορισμών δεν είναι σε θέση να βρουν κατοικία υπό τους όρους της αγοράς. Άρα τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίσουν ομάδες στόχους για την κοινωνική κατοικία και να κατανέμουν την κοινωνική κατοικία με διαφανή τρόπο και ε, κατά προϊόντα σε αυτού που κινδυνεύουν περισσότερο από αποκλεισμό. Τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλο περιθώριο λιγμών για τον καθορισμό του μεγέθου τη ομάδα στόχο. Ο ρόλος της Κομισιόν περιορίζεται στο να ελέγξει ότι δεν υπάρχουν ε, έκδηλα λάθη στους ορισμούς αυτούς. Αυτή η θέση επιβεβαιώθηκε στην απόφαση της Κομισιόν του Δεκεμβρίου του 2009 σχετικά με την κοινωνική κατοικία στην Ολλανδία. Η προσέγγιση αυτή επίσης είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το άρθρο 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που αναφέρεται ε, στην κοινωνική και στεγαστική ε, αρρωγή για όλους αυτούς που δεν έχουν επαρκείς πόρους. Ένας σαφής ορισμό κανονισμός της κοινωνικής επίση επίσης εξασφαλίζει ότι οι κρατικέ ενισχύσει δεν μπορούν να διοχερευτούν σε ε, οικονομικέ και εμπορικέ δραστηριότητε, πέρα από την ε, εμβέλεια τη ε, υπηρεσία δημοσίου ενδιαφέροντο. Όπως είπα, δεν μιλάμε γενικά για στέγη αλλά για κοινωνική κατοικία. Ε, σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας και κατανομής τη κοινωνική κατοικία είναι προ το συμφέρον των ίδιων των δικαιούχων και εξασφαλίζουν σωστή χρήση των δημοσίων κονδυλίων. Απαντώντας τώρα στην ερώτηση υπαριθμών 3, δηλαδή γιατί περιορίζεται η πρόσβαση σε ε, νοικοκυριά με όριο 33.000 ευρώ να ε, αναφερθώ σαφώς στο εξής. Δεν υπάρχει τέτοιο όριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόσβαση σε κοινωνική κατοικία. Αυτό το όριο αφορά μόνο μία χώρα, την, ε, τις κάτω χώρες. και είναι κάτι που αποφάσισαν ε, οι αρχές της χώρας αυτής για να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες για τη γενική ατυχία με τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με, την, ε, ε, με τις κρατικές ενισχύσεις η Κομισιόν δεν βρήκε κανένα λάθος στον ορισμό αυτό για την κοινωνική κατοικία και γι' αυτό ενέκρινε το Ολλανδικό Σχήμα Κρατικών Ενισχύσεων. Ήθελα να πω ότι η ομάδα στόχος αποσορίστηκε από ε, τις Ολλανδικές Αρχές είναι πολύ ε, πλατιά και καλύπτει 33% του Ολλανδικού πληθυσμού. Το λόγο μιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριο Βαν για δύο λεπτά παρακαλώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς τη στιγμή της κρίσης και της συζήτησης που κάνουμε για το πώς θα έχουμε μια βιώσιμη κοινωνία με ανταγωνιστικότητα, ερχόμαστε να συζητήσουμε για κάτι που μπορεί να σας φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά αγγίζει τον πυρήνα ε, των ανησυχιών πολλών. Δηλαδή, ποιος θα πάρει κοινωνική κατοικία. Ακριβώς σε μια περίοδο που οι τράπεζες είναι πολύ πιο επιφυλακτικές από τότε που άρχισε η συζήτηση στην Ολλανδία το 2005 ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση και τώρα οι τράπεζες δεν δανείζουν. Πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα πραγματικό. Και ε, η οροφή των 33.000 ευρώ ε, θα υποβληθεί και στη Βουλή της Ολλανδίας που πρέπει να συμφωνήσει βέβαια ε, με την πρόταση αυτή αλλά 40.000 είναι ε, το όριο, η οροφή για την κοινωνική ασφάλιση. Κανονικά εκεί θα πρέπει να ανεβεί ε, το ποσό. Και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει δυνατότητα ευελιξία στα κράτη-μέλη. Ε, θα πρέπει να έχουν αυτό το περιθώριο. Το 10% είναι χαμηλό ποσοστό. Και εγώ όταν τελείωσα τις σπουδέ μου είχα ένα περισσότερο εισόδημα, αλλά μπόρεσα να μείνω σε μια κοινωνική κατοικία μέχρι να βρω ένα άλλο σπίτι και να μετακομίσω. Να πρέπει να υπάρχει λοιπόν αυτή η ευελιξία. Ε, και σε ό,τι με αφορά εμένα, το συμπέρασμα είναι η επικουρικότητα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που μπορούν να ρυθμίσουν ε, τα πράγματα μόνες τους σε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο και δεν λαμβάνεται παρκώς υπόψη αρχή της επικουρικότητας. Τώρα θα πρέπει να έρχεται ένα ψήφισμα που να απαντά ε, σε αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικά έχει θετική στάση, αλλά ας μην περιορίζει τόσο πολύ τα κράτη-μέλη. Και ο κόσμος εξαρτάται από αυτές τις ρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για την ομάδα ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Γκέμπαρτ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ακούω τη συζήτηση και διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόσετε το δίκαιο στους τομείς αυτούς. Και εσείς κύριε Άντορ είπατε ότι δεν υπάρχει ρύθμιση ευρωπαϊκή που βάζει οροφή 33.000 ευρώ. Οι Ολλανδοί συνάδελφοι λένε βεβαίως υπάρχει ρύθμιση. Ε, έχει ε, γίνει στη χώρα μας ακριβώς. Γιατί φοβηθήκατε ή φοβήθηκαν οι Ολλανδοί ότι αν δεν βάλουν αυτή την οροφή θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τους πει πού είναι τα κριτήρια και επιλεξικότητα. Λοιπόν, γιατί επικρατεί αυτή η ανασφάλεια ακριβώς επειδή είναι πάρα πολλές δυσκολίες στα κράτη-μέλη τα ίδια. Να πάρουν μόνα τους την απόφαση με ε, πνεύμα κοινωνικό και Ε, χωρίς αναλγησία για να μπορεί ο κόσμος να βρίσκει κοινωνική κατοικία όταν τη χρειάζεται. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο που να παρέχει ασφάλεια δικαίου και να ε, ξεκαθαρίζουμε τι επιτρέπεται και τι είναι δυνατό. Γενικά ότι αυτό θα πρέπει να είναι στο γενικό οικονομικό ε, συμφέρον, ότι είναι κοινοφελείς υπηρεσίες αυτές που χρειάζονται προστασία και στα κράτη-μέλη ρυθμίζονται σε τοπικό επίπεδο και είναι καθολικές υπηρεσίες, θα πρέπει όλοι να έχουν... Ε, είχα δύο λεπτά. Ε, είναι καθολικές υπηρεσίες και να φροντίσουμε πραγματικά να προσφέρονται σε όλους τους δικαιούχους. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να το σκεφτούμε και ξέρω ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, υπάρχει ένας προβληματισμός για το πώς θα δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των κοινοφιλών υπηρεσιών, ιδιαίτερα των κοινωνικών. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι τέτοιο πρέπει να το ζητήσουμε και είναι καλό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέμπαρτ. Μένα στον κατάλογό μου έχετε 1,5 λεπτό, αλλά ούτως ή άλλως ξεπεράσατε και τα δύο. Ε, η κυρία Ντυρόν, η αντιπρόεδρος για την ομάδα των Πρασίνων. Madame la Présidente, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εδώ γίνεται λόγος για νομική βάση. Φυσικά και είναι σημαντικό αυτό. Πίσω όμως από την νομική βάση θα ήθελα εγώ να τονίσω το γεγονός ότι η κατοικία και η κοινωνική κατοικία δεν είναι προφανώ μια αγορά ή μια εμπορική δραστηριότητα όπως οποιαδήποτε άλλη. Η κοινωνική κατοικία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εμπορικη δραστηριοτητα οπω οποιαδηποτε αλλη η κατοικία, ε, στέγαση για ανθρώπους με χαμηλά εισόδημα. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα κοινωνική ανάμειξη κτλ. για τα οποία μιλήσαμε, αλλά ε, και κοινωνικές κατοικίες, αυτοί που διαμένουν στις ε, περιοχές ε, ή στις πόλεις ή στην περιφέρεια των πόλεων. Συνδέεται επίσης με ένα ολόκληρο έργο που έχει να κάνει με τους ενίκους, με την αλληλεγγύη των ανθρώπων που διαμένουν σε αυτές τις κατοικίες, σε αυτές τις περιοχές και γι' αυτό θα πρέπει να θεωρείται ως κάτι διαφορετικό Επίση, επειδή θα εργαστούμε και για τα θέματα των υπηρεσιών γενικού συμφέροντο, νομίζω ότι είναι πολύ κακό μήνυμα εδώ να ερχόμαστε και να ε, επισημαίνουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ή τι ενισχύσει για την κοινωνική κατοικία. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, αυτό το όριο των 33.000 ευρώ, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν μονογονεϊκέ οικογένειε, ηλικιωμένοι, ε, κάποιε ε, οικογένειε διαλυμένε ή αναδιοργανωμένε κτλ. Υπάρχουν τέτοια θέματα που ε, θα πρέπει να διέπονται από ευελιξία για να έχουμε πραγματικά κοινωνική κοινωνικές παροχές. Κύριος Λεϊαρίκ, για ένα λεπτό. Κρατήστε το χρόνο που σας έχει παραχωρήσει η πολιτική σας ομάδα, σα παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μόλι είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, προσδώσει μεγάλη σημασία στην κοινωνική κατοικία. Πράγματι, πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο δεν εφαρμόζεται στα κράτη μας. Αυτό λοιπόν είναι ακόμη ένα ε, στίγμα μελανό, μια κοιλίδα μελανή ε, σε, αυτό, σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Επίσης αναφέρατε κάποια συνήθη λόγια ε, της Κομισιόν, όμως η πραγματικότητα που βλέπουμε από την εμπειρία μας είναι ότι ε, η Επιτροπή και το Δικαστήριο ουσιαστικά επαγορεύουν το δίκαιο με βάση μια αρχή καταδικαστική που είναι ο ελεύθερος ε, ανταγωνισμός ε, χωρίς τρευλώσεις που τελικά δημιουργεί προβλήματα στην πρόσβαση στην κατοικία και στην κοινωνική κατοικία. Και ακόμη χειρότερα, το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την κοινωνική κατοικία μόνο για τα άτομα τα οποία ε, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Άρα ουσιαστικά δημιουργεί ένα είδος ε, γκέτου ε, και είναι κατά της ανάμειξης των πληθυσμών σε, αυτά τα, σε αυτές τις κατοικίες. Νομίζω λοιπόν ότι η ίδια αρχή του ανταγωνισμού η οποία γράφεται στις συνθήκες είναι αυτή που θα πρέπει να αλλάξει. Ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε. Από την άλλη πλευρά λοιπόν φοβούμε ότι οι δηλώσεις του Πρόεδρου Μπαρόζο που επιβεβαίωσε το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ σήμερα που μάλλον ουσιαστικά θα οδηγήσουν σε έλεγχο των προπολογισμών, θα μειώσουν τι δαπάνε για τι εργατικέ κατοικίε και ιδίω για τι κοινωνικέ κατοικίε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει σε νέε βάσει πλέον να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ συγγνώμη, λέει στα γαλλικά η πρόεδρο, αλλά ε, ξεπεράσει το χρόνο γόρευσή σα και αυτό είναι άδικο για του συναδέλφου. Η πολιτική σα ομάδα σα δίνει περισσότερο χρόνο τον κατάλογο των άλλων ομιλητών. Σας παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Είναι αργά, πρέπει να τελειώσουμε στην ώρα μας. Ο κύριος ε, Έγγελ έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω κάπως με την Ιζαβέλ Ντουιράν, που σωστά είπε ότι η κοινωνικές κατοικίες δεν είναι εμπορικός τομέας που θα πρέπει να είναι στην ανταγωνιστικότητα όπως όλοι οι άλλοι τομείς οικονομίας. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει και ο κύριος Επίτροπος. Αυτό που διακυβεύεται είναι κρατικές ενισχύσεις. Μα πώς είναι δυνατόν, διερωτώ με. Αφού είναι κοινωνική ε, παροχή, δεν θα υπάρχει ε, κρατική ενίσχυση προς τους δικαιούχους και ε, προς τις ε, ε, εταιρείε και τις φορείς που διαχειρίζονται βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Δεν στρεβλώνουμε τον ανταγωνισμό έτσι. Εγώ βέβαια θα μιλήσω μόνο βάσει της δικής μου εμπειρίας στη χώρα μου. Οι κοινωνικές κατοικίες παρέχονται με πολύ διαφορετικά κριτήρια και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να μας ορίσει μέχρι τελευταία τελείας ποιο πολίτη, θα πρέπει να δικαιούται τη κοινωνική στέγη και με ποια κριτήρια και με ποιε προϋποθέσεις. Μπορεί να διαφέρει η κατάσταση ακόμα και από τόπο σε τόπο ή από την εξέλιξη της οικογένειακή κατάσταση κάποιου που μπορεί να ζούσε στο παρελθόν με την οικογένειά του, τα χωρίς την οικογένειά του ε, το εισόδημα κυμαίνεται, όπως είπε και ο κύριος Βανίσεροι Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου δεν έχει πάντα το ίδιο εισόδημα. Μπορεί μια μέρα να δικαιούται κοινωνική κατοικία με κάποια κριτήρια και αργότερα να ε, του αφαιρείται το δικαίωμα αυτό. Τώρα δεν ξέρω, αυτά που ζητάτε ε, δεν μου φαίνονται σωστά. Δεν θα πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερβεί τον εαυτό τη για να μα ε, επιβάλλει ή να μας προτείνει, εν περιπτώσει, αλλά μας επιβάλλει κανόνες ε, που δεν μας επιτρέπουν την ευελιξία και είναι και ανάλγητε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ονζέλ. Τώρα ε, ο κύριο Ντεγόσα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμμετείχα στη συζήτηση αυτή ω εισηγητή τη Επιτροπή Απασχόληση για το μέλλον ε, των υπηρεσιών γενικού συμφέροντο. Το όλο αυτό θέμα ε, φαίνεται να σχετίζεται με το σοβαρό πρόβλημα της παροχής κοινωνικής κατοικίας για τους πολίτες και τη σχετική απόφαση της Κομισιόν. Λυπάμαι που η Κομισιόν δεν έχει δεν προτίθεται να υποβάλει ε, άλλες σχετικές προτάσεις πέραν του ισχύοντος συστήματος. Ε, καλό την Κομισιόν να δημιουργήσει νομική βεβαιότητα και σαφήνεια ε, για τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για τις υπάρχουσες υπηρεσίες, ιδίω τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και για να καλυφθούν νέες κοινωνικές ανάγκες. Διότι όχι μόνο πρέπει να έχουν οι πολίτες ένα δίκτυο ασφαλείας σε περίπτωση ανάγκης, αλλά να υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο να εξυπηρετεί όλους τους πολίτες. Η υγεία, η στέγη και η παιδεία είναι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται σε καθολική βάση και όχι μόνο ε, σύμφωνα με τις ε, ε, ανάγκες της αγοράς. Η καθολικότητα και η ε, ανάγκη ποιότητας στους τομείς αυτούς είναι κάτι το προφανές. Πρέπει να παρέχεται ε, μέσα από τα στήματα αυτά μια κοινωνική αξία που δεν μετρέται σε κανένα οικονομικό ισοζύγιο και πέρα από τις πιέσεις της αγοράς. Οι σημερινές ανεπάρκειες πρέπει να καλυφθούν και σε εθνικό και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διότι οι ανισότητες αυτές δεν μπορούν να συνεχιστούν περαιτέρω. Madame le Président, chers collègues. Κυρία... Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, πρώτα απ' όλα μια διαπίστωση δεν υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα στα θέματα της πολιτικής ε, κατοικίας και ιδιαίτερα της κοινωνικής κατοικίας. Παρ' όλα αυτά, στην απόφαση την οποία αναφέρουμε σε αυτή την προφορική ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έναν ορισμό της κοινωνικής κατοικίας. Και αυτό αναφέρθηκε πολλές φορές. Το πρόβλημα της κοινωνικής κατοικίας και της πρόσβασης στη στέγη σήμερα σε περίοδο κρίσης είναι ένα μείζον πρόβλημα, κύριε Επίτροπε. Ας ξαναβάλουμε λίγη ανθρωπιά σε όλες αυτές τις τεχνικές, νομικές, τεχνοκρατικές συζητήσεις μας. Πέρα από τη στέγη καθ' αυτή, η κοινωνική κατοικία είναι το θεμέλιο μιας πραγματικής ένταξης, μια πραγματικής ενσωμάτωσης στην κοινωνία για αυτούς που επωφελούνται. Ο ορισμός που διώθηκε στα πλαίσια του ελέγχου ε, των κρατικών ενισχύσεων εκ μέρους της Κομισιόν είναι εντελώς ε, αμφισβητήσιμος. Ο Δεκάρτ, ο Καρτάσιος, ο μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος που γεννήθηκε στην περιοχή μου, στο Λίγυρα, ε, είπε ότι το γενικό συμφέρον είναι ένας κύκλος που ξέρουμε το κέντρο του, αλλά όχι την περιφέρειά του, κύριε πίτροπε Σας θέτω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Πρώτη απλή ερώτηση. Ποια είναι η νομική αξία ενός τέτοιου ορισμού. Και ε, υποτίθεται ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Η δεύτερη ερώτηση είναι πολύ πιο γενική. Κατά την άποψη της Κομισιόν, πού ξεκινάει και πού σταματάει η κοινοτική αρμοδιότητα ε, σχετικά με την οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών. Γιατί το ερώτημα αυτό είναι τελικά σημαντικό. Έχει να κάνει με την καθολικότητα και την προσβασιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Σιμών έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, παντού στην Ευρώπη οι Δήμοι και οι κοινότητε μας έχουν προβληματικέ συνοικίε. Παντού προσπαθούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, ακριβώ όταν είναι μειονεκτικές συνοικίε. ε, να προσπαθήσουμε να φέρουμε τις συνοικίες και τον κόσμο πιο κοντά στην κανονική ζωή της πόλης. Έχουμε κριτήρια για τις κοινωνικές κατοικίες, ε, ε, αλλά κριτήρια τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Αυτό ε, αποκλεί, ε, αν βάλουμε αυτά τα κριτήρια, την οποιαδήποτε ανάμειξη των κοινωνικών ομάδων και του πληθυσμού. Και αυτό έρχεται να καταρρύψει όλες τις προσπάθειες και να καταστρέψει όλες τις προσπάθειες δεκαετιών ε, των Δήμων και κοινοτήτων. Και αυτά τα έχει ζητήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινοτική πρωτοβουλία Urban 1 και 2. Ποια είναι τα κριτήρια για την κοινωνική στέγη, αν τα περιορίσουμε μόνο αποκλειστικά στους πιο φτωχούς, τους πιο ενδεείς, τους πιο ε, ανεκτούντες ε, πολίτες και να το θεωρήσουμε ότι είναι επιδότηση, τότε ακριβώς αποτρέπουμε αυτή ε, την ανάμιξη του πληθυσμού, του να ζει ε, ε, ο κόσμος και ε, στις μειονεκτικές ε, περιοχές μαζί. Και τελικά έχουμε κοινωνικό αποκλεισμό και αυξάνουμε τα προβλήματα και τα μεγεθύνουμε στις πόλεις μας. Γι' αυτό χρειάζεται ευρύ ορισμός και ευρύ αρμηνία της αρχής της επικουρικότητας. Και θα ευγνωμονούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μας απαντούσε από αυτού. Ευχαριστώ. Σύντομα. Ο κύριος Ζέλερ τώρα για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι τώρα το ερώτημα για την αρχή της επικουρικότητας και της καθολικότητας των κοινοφιλών υπηρεσιών γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στο παράδειγμα της Ολλανδίας βλέπουμε την κοινωνική κατοικία τώρα να ε, κυριαρχεί στη συζήτηση. Δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση αυτό. Χρόνια ολόκληρα οργανώσεις ενοικιαστών και εκπρόσωποι τους ε, υποπτεύονται ότι η πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα στραφεί, θα περιορίσει την κοινωνική κατοικία. Μέχρι και ε, θα την καταστρέψει τελείως φοβούνται. Ε, μετά από την τροφή και την ένδυση, βασική ανάγκη του ανθρώπου είναι η στέγη. Και είναι κοινωνικό αγαθό. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε την ύπαρξη αστέγων στις πόλεις μας. Είναι κοινωνική πρόκληση. Έτσι λοιπόν, Υπάρχουν κράτη που ενδιαφέρονται για την ευημερία των πολιτών τους και ενισχύουν την κατοικία ή υποστηρίζουν ε, τους πολίτες στην αγορά στέγης. Τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα ιδιαίτερο περιστατικό μετά την ένταξη πολλών ε, χωρών της Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Επειδή είναι διαφορετική η δομή ολόκληρη της κατοικίας και της στέγης στην ε, Ανατολική Ευρώπη ε, χρειάζεται κάπως να είναι συγκρίσιμες οι δομές ε, της κοινωνικής στέγης και της ενίσχυσης της κατοικίας. Σε πολλέ χώρε τη Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη ιδιωτικοποιήθηκε η στέγη μετά την πολιτική αλλαγή που έζησαν οι πολίτε Και γιατί δεν υπήρχε και επαρκής κατοικία. Ε, αντέδρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενέκρινε διαρθρωτικά κονδύλια για τις στέγη της χώρας αυτές. Παρ' όλα αυτά όμως η πολιτική ε, της ε, κατοικίας είναι ένα θέμα που αφορά τα κράτη-μέλη της περιφέρειας και ιδιαίτερα τους δήμους και κοινότητες. Είναι κλασική περίπτωση επικουρικότητας. Δεν μπορεί να ρυθμίζεται, ούτε χρειάζεται υπερεθνική ρύθμιση. Και το κοινωνικό αγαθό ακριβώς είναι ένα ε, αγαθό και δεν ε, ισχύει η αγορά εδώ. Η κυρία Γοηνιέ έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Respectez le temps de parole, Madame Vorsitzende. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Κοινοφιλείς υπηρεσίες και κοινωνικές υπηρεσίες ε, ε, ενισχύονται ε, γνωρίζουμε άλλα μεγάλες δυσκολίες και οικονομικές και διαρθρωτικές, οι οποίες δυσκολίες ενισχύονται ακριβώς από την κοινωνική και την οικονομική κρίση. Αλλά σε καιρούς ανασφάλειας, ε, οικονομικής κρίσης ε, και άγχους για το μέλλον, οι κοινωνικοί σταθεροποιητές είναι σημαντικότεροι από ποτέ. Εγώ είμαι από τη Βιέννη και υπάρχει η βασική ιδέα της κοινωνικής κατοικίας που σημαίνει φθηνή, ε, κατοικία για ευραία στρώματα του πληθυσμού και όπως, όχι όπως το ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, πολίτες που είναι ε, οικονομικά ασθενείς ή μειονεκτούντες γιατί αυτό δημιουργεί γκέτο. Δεν σας κρύβω την απόψή μου ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, δικαίωμα και αρχή ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρέχει κοινοφελείς υπηρεσίες και κοινωνική κατοικία και να, κάνει, ε, να ορίζει μάλλον η ίδια η τοπική αρχή ποια είναι η κοινωνική κατοικία και ποια είναι τα κριτήρια. Οπωσδήποτε όμως αυτό που χρειάζεται είναι ασφάλεια δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφήνεια και νομικά εργαλεία έτσι ώστε οι κοινοφελείς υπηρεσίες να είναι καλά ορισμένες. Η, κυρία Κέλλη έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, ε, ε, Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που διευκρίνησε ορισμένα σημεία που τέθηκαν με την προφορική ερώτηση και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η παροχή στέγης είναι απόλυτη αναγκαιότητα για οποιονδήποτε. Ιδίω ε, στις σύγχρονες κοινωνίες ε, πρέπει κάποιος να έχει τη σκεπή πάνω από το κεφάλι του. Αυτό είναι ένα δικαίωμα για όλους και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι αυτό θα πρέπει ε, να παρέχεται με δικά μας μέσα ή μάλλον να παρέχει τη στέγη ο άνθρωπος είτε με τα δικά του μέσα είτε με τη βοήθεια της κυβέρνησης των υπηρεσιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την παρέμβαση ε, μιας χώρας συγκεκριμένη, σε ό,τι αφορά την κοινωνική κατοικία, έχω να πω ότι στη δική μου χώρα υπήρξαν φορολογικά κίνητρα που οδήγησαν τελικά στο να σκάσει φούσκα στα κίνητα, να σκάσει στην υποδομή. Υπήρξαν... Ε, ε, κάποιες απαλωτριώσεις και κάποιες άλλες εξελίξεις για τη δημιουργία κατοικίας λόγω φορολικών κινήτρων. Δόθηκαν ε, γενναιόδωρα δάνεια σε εργολάβους που μετά δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν. Δόθηκαν επίσης δάνεια σε πολίτες για να αγοράσουν σπίτια που δεν μπορούσαν ούτε αυτοί να τα αποπληρώσουν και έτσι έσκασε η φούσκο, όπως σας είπα. Θα πρέπει λοιπόν γενικώ και το κράτο ε, να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτόν τον τομέα. Αλλά η παροχή κοινωνική κατοικία σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα το ότι βασίζεται στο εισόδημα, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα περιοριστική και δεν έχει και νόημα. Και ακούσαμε λόγους από πολλούς προλαλήσαντες. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ευρύτερη έννοια ίσως καλό θα ήταν να δώσει κάποιε κατευθυντήριε γραμμές, να βοηθήσει για την παροχή κοινωνικής κατοικίας, αλλά όχι να είναι ιδιαίτερα ε, υπαγορευτική και περιοριστική σε ό,τι αφορά όρια για εισόδημα κτλ. Αυτό δεν έχει νόημα δεν θα έχει αποτέλεσμα και δεν θα πρέπει να επιχειρηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη, ακριβής και στον χρόνο σας. Η κυρία Τιτσάου για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η κοινωνική κατοικία, κατοικία ανήκει στις υπηρεσίες γενικού Συμφέροντο. Δυστυχώ, σήμερα η ανεργία φτάνει το 20% στους νέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες υπάρχει μια ποσόστοση της τάξης του 4% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κράτη-μέλη για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και για την ενεργειακή απόδοση των κτίριων. Ωστόσο, και δυστυχώς λόγω της οικονομικής κρίσης, η οικονομική κατάσταση των οικογενειών στην Ευρώπη επιδεινώνεται και η πολύ υψηλή μεταξύ των νέων ανεργία είναι κάτι που μας ανησυχεί. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Επίτροπε, σας ζητούμε να μας βοηθήσετε. Να εξασφαλίσετε δηλαδή ότι για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, δημοσιονομικού προγραμματισμού, αυτή η ποσόστοση για την ενεργειακή απόδοση των κτίριων και την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών να αυξηθεί και να φτάσει στο 15%. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε την απαιτούμενη σημασία στην κοινωνική κατοικία και στου νέου και στου ηλικιωμένου. Αυτέ οι δημόσιε υπηρεσίε είναι πολύ σημαντικέ για την προστασία, για την ένταξη όλων των πολιτών στην κοινωνία. Υπό τον όρο βέβαια ότι θα είναι προσβάσιμε για όλου του πολίτε αυτέ οι υπηρεσίε. Για να αποτελέσει αυτό λοιπόν πραγματικότητα σε όλα τα κράτη-μέλη, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει μια οδηγία πλαίσιο για τι δημόσιε υπηρεσίε όπου θα θεσπίζονται ε, κατώτατοι κανόνες και προϋποθέσεις και θα εγγυάται αυτός ο κανονισμός την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών, θα εγγυάται επίσης την ποιότητα και την ε, διαφάνεια. Ο κύριος Κορέρα Ντεκάμπος, για ένα λεπτό παρακαλώ. Senhora Presidente, Senhor Comissário, a habitação social é um serviço económico de interesse geral. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η κοινωνική κατοικία είναι μια υπηρεσία γενικού συμφέροντος και ε, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για τις αγορές και για την κοινωνία. Το άρθρο 26 του πρωτοκόλλου της Συνθήκης της ε, Λισαβόνας αναφέρει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι αρμόδιες για την παροχή αυτού του είδους ε, της υπηρεσίας. Γι' αυτό ο περιορισμός της ομάδας στόχου σε νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των 33.000 ευρώ είναι κάτι που δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Αυτό αυτό είναι ένα καθαρά οικονομικός ορισμός της φτώχεια και δεν λαμβάνει υπόψη την επικοινομορφία των 27 ε, κρατών μελών. Δεν είναι καθαρά θέμα φερεγγιότητας, οικονομικής ευχέρειας. Η κοινωνική κατοικία αφορά και κοινωνικούς και πολιτιστικούς ε, λόγους, ε, ε, λόγους που έχουν να κάνουν με την εργασία, με την κοινικότητα των γυναικών, την κοινικότητα των πολιτών μέσα στην Ευρώπη και ο αγώνας που δίνουμε για να φύγουμε από την οικονομική κρίση σημαίνει ότι χρειαζόμαστε την οικονομική ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερη μετανάστευση, μεγαλύτερη πολιτισμική ποικιλομορφία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπορέσουν να ενταχθούν, να ε, καταπολεμηθεί η περιθωριοποίησή τους. Ε, μήπως η Κομισιόν μπαίνει εδώ σε χωράφια που ανήκουν στα κράτη-μέλη. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της ε, διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας στις ε, κοινωνικές υπηρεσίες και το ρόλο που έχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Τα θέματα της κοινωνικής κατοικίας έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος και η αλήθεια είναι ότι η κρίση άφησε πολλούς εργαζόμενους με την ανάγκη για κοινωνική κατοικία. Αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά πρότυπα ε, όταν αποφασίζουν σχετικά με τα κριτήρια για την κοινωνική κατοικία. Είναι κατανοητό ότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Για να εφαρμοστεί το δικαίωμα ε, πρόσβασης στις καθολικές υπηρεσίες, πιστεύω ότι είναι λογικό να οριστούν κάποιες γενικές αρχές και να καθοριστεί ένα ανώτατο εισόδημα ε, σαν σύσταση σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως τη διακριτική ευχαίρεια για τη λήψη των αποφάσεων θα πρέπει να την τα κράτη-μέλη να βάζουν υπόψη κοινωνικές και οικονομικές διαφορές. Ευχαριστώ. Στη διαδικασία Catch the Eye θα πάρουν το, το, το λόγο οι συνάδελφοι για ένα λεπτό. Ο κύριος Νικολέσκου πρώτος. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Επίτροπο για τις διευκρινήσεις του σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Ούτε εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ενιαίο ορισμό για τις κοινωνικές κατοικίες. Είναι δύσκολο να έχουμε μια ομοιόμορφη ρύθμιση σε όλα τα κράτη-μέλη γιατί έχουμε διαφορές και διαφορές στο βιωτικό επίπεδο. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το θέμα της επικουρικότητας. Επιτρέψτε μου να ξεφύγω λίγο από το αυστηρό πλαίσιο της ερώτησης. Ε, θα πρέπει να έχουμε πιο ξεκάθαρες προδιαγραφές ε, και κριτήρια στην επιλεξιμότητα των κοινωνικών κατοικιών για κοινότητες περιθωριοποιημένες. Ε, το Φλεβάρι, ενέκρινε έκθεση ναι, ναι, στο Κοινοβούλιο, το ανέφερε και η κυρία Τσικάου αυτό και θα ήθελα να σας πω ότι καλό θα ήταν να αυξηθούν τα κονδύλια που δίνονται. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Νταρντάν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ανησυχώ και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, πολλοί περιφέρειες στην Ευρώπη, όπως η δική μου, ε, αυτό το καιρό θέλουν να μεταρρυθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο χορηγούν τις ε, κοινωνικές κατοικίες για να αποφύγουμε τα γκέτο και τη συνένωση ε, μειονεκτούν των πληθυσμών στα ίδια κτίρια και στις ίδιες συνοικίες. Η απόφασή σας αντιτίθεται στην απαραίτητη κοινωνική ανάμειξη και εξισορρόπηση. Δεν είναι σωστό, κύριε Επίτροπε, να εμποδίζονται τα κράτη-μέλη να ασκούν αυτή την πολιτική. Βεβαίω, οι γενικέ υπηρεσίε, κοινοφελεί υπηρεσίε για τη στέγη ε, μπορούν να έχουν κριτήρια ε, για συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά να μπορούν τα κράτη-μέλη να ορίζουν ε, τα κριτήρια αυτά και πώς θα αναμειγνύεται ο πληθυσμός στις συνοικίες και στις γειτονιές θα πρέπει με τα ίδια τα κράτη-μέλη, τι περιφέρειε και τους ΟΤΑ να γίνεται αυτό, όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι το δικαίωμα στην στέγη, στην κατοικία είναι ένα θεμελιώδε δικαίωμα. Κατά συνέπεια, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποχρέωση να εγγυηθούν την κοινωνική κατοικία σε όλα τα άτομα που νιώθουν την ανάγκη αυτή. Σε στιγμέ ε, βαθιά ε, κοινωνική κρίση, όπου ο αριθμό των ατόμων και των οικογενειών που είναι πολύ χρεωμένε ε, και έχουν μεγάλε δυσκολίε στο να τα βγάλουν πέρα, να πληρώσουν το ενίκιο τους, παραδείγματο χάρη, το σπίτι τους, το διαμέρισμά τους. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο ε, να υποστηρίξουμε τις οικογένειες που δεν έχουν τους απαραίτητους σπόρους να έχουν μια αξιοπρεπή κατοικία με τις απαραίτητες υπηρεσίες, με τις κατάλληλε υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να μπορέσουν να ε, χρησιμοποιήσουν ε, ε, οι κυβερνήσεις, τα κράτη, τα προβλεπόμενα κονδύλια για να εγγυηθούν την κοινωνική κατοικία, στην οποία έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες και να θέσουν ένα τέρμα στις κοινωνικές ανισότητες και να ευνοήσουν την κοινωνική ένταξη. Καλό θα ήταν λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει προς, ε, προς την κατεύθυνση αυτή, χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο την αρχή της επικουρικότητας και υποστηρίζοντας την καθολικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών. Ε, η κυρία Ζαμπόρσκα έχει το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ.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 το πρόβλημα είναι ότι οι ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν διαστρεβλώσει την κατάσταση στην αγορά και τον ορισμό της κοινωνικής κατοικίας. Ε, ε, το θέμα είναι ότι η κοινωνική κατοικία εξαιρείται από την υποχρέωση κοινοποίηση για τις κρατικές ενισχύσεις ε, και έτσι η αρμοδιότητα βρίσκεται πλήρως στα χέρια των εθνικών αρχών και των τοπικών ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, δεν θα πρέπει να αμφισβητούμε την ικανότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα την κατάσταση και είναι σε θέση να λύνουν τα προβλήματα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, panie komisarzu, otóż... και κύριοι, ε, κύριε Επίτροπε, μπορούμε να δούμε πολύ καθαρά ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει διαφορετική όψη στα διάφορα κράτη-μέλη. Στην Πολωνία έχουμε διάφορες περιφέρειες όπου ε, υπάρχουν πολλοί άστεγοι λόγω του χαμηλού εισοδήματός τους. Συνήθως είναι οι τοπικές αρχές αυτές που ε, ασχολούνται με τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Η δουλειά του είναι να παρέχουν βοήθεια όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Χωρίς την υποστήριξη των τοπικών αρχών, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα είχαν κανένας είδους υποστήριξη και βοήθεια. Αν ε, πρόκειται να εφαρμόσουμε ε, έναν εναρμονισμένο ορισμό στις σχετικές πολιτικές, πρέπει να σκεφτούμε πώς στο μέλλον θα ήταν δυνατόν να χορηγηθούν επιπλέον κονδύλια στις τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλίσουν την κοινωνική κατοικία που είναι τόσο απαραίτητη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριο Σάντερ. You have the floor, Mr. Commissioner. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, ε, συμφωνώ απολύτω ότι πρέπει να δούμε το θέμα αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο πλαίσιο συγκεκριμένα τη ε, χρηματοπιστωτική και οικονομική ε, κρίση. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε ένα τεστ για τι πολιτικέ ανταγωνισμού στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στον τομέα των αυτοκινήτων ή και στον τομέα τη στέγη. Ήταν επίση ένα τεστ και για τι κοινωνικέ μα πολιτικέ. Είτε αυτέ αφορούσαν τα παιδιά, είτε του ηλικιωμένου, είτε του άστεγου. Και ε, στα πλαίσια αυτού του συνόλου ερωτήσεων που έλαβα, αυτά τα δύο θέματα, ο ανταγωνισμός δηλαδή και οι κοινωνικές πολιτικές, επικαλύπτονται και γι' αυτό το θέμα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο ε, από ό,τι θα ήταν ε, έξω από τις συνθήκες κρίσης. Η κρίση έδειξε ένα μια τεράστια έλλειψη ε, της αγοράς ε, και στον τομέα της στέγης, όχι μόνο στο χρηματοπιστωτικό ε, τομέα. Και αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν μπορούν να λύσουν αυτά τα προβλήματα, όχι μόνο για τους ε, πολύ φτωχούς, αλλά και για ευρύτερε ομάδες της κοινωνίας. Και γι' αυτό είμαι σαφώς εναντίον οποιασδήποτε αρχής που θα περιόριζε την έννοια της κοινωνικής κατοικίας μόνο για τα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας. Και ιδιαίτερα, ε, αν λάβουμε υπόψη μας την ε, ποικιλομορφία των ε, κοινοτικών χωρών και την αρχή της επικουρικότητας, σίγουρα θα έπρεπε να αφήσουμε τους σχετικούς ορισμούς στα ίδια τα κράτη-μέλη, όπως είπα ήδη στις αρχικές μου απαντήσεις. Επανερχόμενος τώρα στο, στην Ολλανδική περίπτωση που είναι η αιστεία όλη αυτή τη συζήτηση, το επίκεντρο τη συζήτηση. Ήθελα να επαναλάβω ότι η Κομισιόν δεν επιβάλλει τα κριτήρια τα οποία θεσπίστηκαν ε, στα πλαίσια τη Ολλανδία και στι άλλε χώρε. Ε, με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας λέμε ότι τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να αποφασίσουν τις συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις για τη χορήγηση κοινωνικής κατοικίας. Και εμείς απλώς επιβεβαιώσαμε την, ε, ε, στην απόφασή μας την ε, έγκριση του Ολλανδικού ε, σχήματος που όπως λέμε καλύπτει με τους ορισμούς ε, το 33% του Ολλανδικού πληθυσμού σίγουρα δηλαδή περισσότερες από τις φτωχότερες απλές ομάδες επιπλέον ε, η Ολλανδική πολιτική εξασφαλίζει την απαραίτητη διαφάνεια και κοινωνική ανάμειξη και δεν περιορίζεται ε, στο να καλύπτει μόνο αυτούς που απειλούνται από ακραίες συνθήκες ε, ένδυας. Ε, ο κίνδυνο τα τελευταία χρόνια αφορά ευρύτερα στρώματα τη κοινωνία, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι πάνω σε αυτό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν ε, ελέγχει μόνο τις ενισχύσεις που δίνονται σε εταιρείε που κατασκευάζουν κατοικίε και όχι σε άμεσες ε, ενισχύσεις προς διάφορα στρώματα του πληθυσμού η Ολλανδική απόφαση ε, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που αφορά γενικότερα τις υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό και να τονίσω ότι πέρα από τη στέγη υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και ιδιαίτερα άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν έναν ε, ρόλο προληπτικό, ένα ρόλο κοινωνικής συνοχής και στοχεύουν σε ολόκληρο το πληθυσμό, ανεξαρτήτως πλούτου ή εισοδηματός. Ε, και αυτό το ξεκαθάρισε η Κομισιόν στην ε, ανακοίνωσή της του 2007 όπου υπογράμμισε τους στόχους και τις προτεραιότητες των ε, κοινωνικών υπηρεσιών. Η Κομισιόν είναι δεσμευμένη στο θέμα της προώθησης της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών. Παραδείγματο χάρη, υποστηρίξαμε την ανάπτυξη ενός, ενός ποιοτικού πλαισίου για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος κάποιες τελικές σκέψεις για να ολοκληρώσω τις απαντήσεις μου. Εφόσον κάποιες από τις ερωτήσεις αφορούσαν ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και τις επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές, θα συμφωνούσα ότι ε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα επηρεαστεί και το θέμα της κατοικίας. Ε, ιδίως σε σχέση με τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν με σκοπό την ε, ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Θα αναπτυχθούν διάφορες δραστηριότητες ε, στον τομέα αυτό, ε, χωρίς βέβαια να επιδιώξουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στέγης. Επίσης, θα υπάρξουν και άλλα θέματα, όπως ε, το θέμα της ε, στέγης για τις πιο ευπαθείς ομάδες ε, του πληθυσμού, όπως για τους Ρώμα. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που έχει ήδη αρχίσει και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξη των διαρθωτικών ταμείων για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της στέγης για αυτές τις ιδιαίτερα ευπαθείς και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες που υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτό όμως ακόμα μια φορά υπογραμμίζει την ε, σημασία του να έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση γιατί οι χώρες πραγματικά διαφέρουν όσον αφορά τις κοινωνικές ανάγκες και σίγουρα οι αποφάσεις ε, και οι λύσεις που εφαρμόζονται σε χώρες υψηλού εισοδήματος δεν πρέπει αναγκαστικά να ακολουθηθούν και σίγουρα δεν πρέπει να επιβληθούν και στα άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έλξε εδώ. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι δήλωση της Επιτροπής με θέμα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.